πώς άρχισε όλη αυτή η ιστορία της εξαφάνισης, ε, θα μπορούσατε ίσως ε, να μας ε, καθησυχάσετε για τα μέτρα που μπορεί να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αποφύγει μελλοντικά τέτοια κρούσματα. πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Ε, για την ε, υποστήριξη του, ε, για την παραγραφή αυτού του ποσού. Πριν από 10 χρόνια συνέβη αυτό και η νομική μας υπηρεσία και η νομική συμβουλή χρειάστηκαν 10 χρόνια για να καλύψουν πώς θα ανακτήσουμε τα ποσά από την τράπεζα. Γιατί η τράπεζα ευθύνεται και πρέπει να εκταμιεύσει το ποσό. Βέβαια είναι ασυνήθιστο γιατί συνήθως ε, υπάρχει μεγάλη προστασία για τις πληρωμές που πρέπει να γίνουν. Μπορώ να το ερευνήσω, δεν είμαι ακριβώς αρμόδιος, αλλά... Τέλος πάντων, μας υποβάλλατε αυτή την ερώτηση επίσημα. Έκτοτε δεν σημειώθηκε τέτοιο κρούσμα, κάνουμε πληρωμές ανά τον κόσμο. Θα μπορούσαμε να το διαβάσουμε στον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή στην Επιτροπή. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάντως ε, ε, συνήθως υπάρχει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας. Οι δικαστές σε αυτή την περίπτωση αποφάσισαν πάντως πως η τράπεζα ε, βάσει της σύμβασης κατέβαλε την πληρωμή και άρα δεν ευθύνονται. Είναι ατυχές βέβαια γιατί πτώχευσε η τράπεζα ε, και υπήρχε και απάτη όμως εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Από τη δική μας οπτική γωνία ε, εξετάζουμε όλες τις πληρωμές ε, για ύποπτες ε, περιπτώσεις στην Αργεντινή πριν από 10 χρόνια εσχάτως με το Αφγανιστάν ή με την Ισλανδική κρίση. Οπότε σταματάμε τις πληρωμές και ερχόμαστε σε επαφή με τους δικαιούχους για να είμαστε σίγουροι ότι μπορούν να τις δεχτούν για να μην δημιουργείται πρόβλημα. Είμαστε σε εγρήγορση πάντοτε ούτως ώστε να έχουμε μία μακροθεώρηση της κατάστασης. Ε, είναι εξαιρετικά περίπλοκο να αποδοθούν ευθύνε πάντως και θα σταματήσω εδώ. Προεδρο, ο κύριος Χάρτον έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ποια μέτρα συγκεκριμένα ανέλαβε για να αποφύγουν μελλοντικά κρούσματα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως μόλις σας είπα, έκτοτε δεν είχαμε κανένα κρούσμα και είμαστε ε, πολύ προσεκτικοί. Εν γέννη υπήρχε ένα τομέα όπου συνήθω υπήρχαν προβλήματα. Όπω σα είπαμε το Αφγανιστάν, μόλι μάθαμε ότι ενδεχομένω θα δημιουργεί το πρόβλημα, ε, σταματήσαμε. Πάυσαμε όλε τι πληρωμέ μέχρι να τι ελέγξουμε μία-μία και να δούμε ποιο εμπλέκεται. Είχαμε επίσης πρόβλημα με την Ισλανδική κρίση, ε, τράπεζες ε, που θεωρούσαμε υγιείς σε διάστημα μίας-δύο ημερών ε, ξαφνικά ασθενούσαν και ερχόμασταν σε επαφή με τους δικαιούχους απευθείας μέσα από τα δίκτυα που έχουμε. Και ξαναλέω πριν από 10 χρόνια συνέβη αυτό, απλώς μας πήρε 10 χρόνια για να διερευνήσουμε την υπόθεση. Ευχαριστώ. Το ελεκτικό συνέδριο είναι παρόν, καταγράφει αυτά που λέμε για αυτή την υπόθεση, την οποία γνωρίζει καλά και γνωρίζετε ότι είμαστε και στην ε, διαδικασία διορισμού ενός νέου διευθυντή της ΟΛΑΦ. Έχουν γίνει προτάσεις από το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν και θα εξεταστούν από το Συμβούλιο και θα πρέπει ίσως να ευαισθητοποιήσουμε το νέο διευθυντή της ΟΛΑΦ σε τέτοιου είδους φαινόμενα και προτείνω, <clears throat> εάν συμφωνείτε, να στείλω και εγώ μια επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου του Προεπολογισμού για να υπενθυμίσω αυτό το λυπηρό επεισόδιο και να παροτρύνω την Επιτροπή Ελέγχου του Προεπολογισμού να είναι ιδιαίτερα επάγρυπνη για τα θέματα αυτά και τέτοιου είδους προβλήματα τα οποία δεν πρέπει να επαναληφθούν. Ωραία. Μετά από αυτές τις διευκρινήσεις, ο εισηγητής μας υποστηρίζει τη μεταφορά. Όχι, κύριε Σουριάν. Ναι, ναι, είναι υπέρ, είναι υπέρ πράγματι. Νόμιζα θέλετε το λόγο. Λοιπόν, ποιος είναι υπέρ αυτής της μεταφοράς. Ευχαριστώ, κατά. Αποχές. Μία αποχή. Η 58 λοιπόν, η μεταφορά 58 έχει εγκριθεί. Κύριε Σιγητά, η 59. στη μεταφορά αυτή μεταφέρονται διοικητικές δαπάνες στη γραμμή ΙΝΤΕΣ όσο μικρότερες οι διοικητικές δαπάνες τόσο το καλύτερο. Αυτή είναι η θέση του Κοινοβουλίου συνολικά. Θα μπορούσαμε να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτή την πρόταση. Αλλά έχω απλώ μια μικρή παρατήρηση ότι συγκεκριμένα αποσύρουμε πάνω από 3 εκατομμύρια από τον εκτελεστικό φορέα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας <clears throat> που θα πάρει πίσω 3 παραπάνω εκατομμύρια στον προϋπολογισμό του 2011. Περικόπτουμε λοιπόν κονδύλια αλλά θα τα επιστρέψουμε αμέσως του χρόνου. Αν δεν χρειάζονται τα λεφτά εφέτος για διοικητικές ε, δαπάνες, Ίσως δεν τις χρειαστούν του χρόνου. Δεν χρειαστούν τα λεφτά για αυτά του χρόνου. Πρέπει να επαφιεθούμε στην σοφία της Κομισιόν και ούτως ή άλλως τα χρήματα έχουν ζητηθεί, επομένως προτείνω να υπερψηφίσουμε αυτή τη μεταφορά. Και να πω επίσης ότι αυτές οι μεταφορές μπορούν να ψηφιστούν και στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Έχουμε αρκετό χρόνο, αλλά εγώ προτείνω να τις ψηφίσουμε τώρα. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι γι' αυτό και κυρίως το ότι εγώ δεν θα μπορώ να είμαι παρόν στις 8 Δεκεμβρίου. Θα ήθελα, αν μπορούμε λοιπόν, να ψηφίσουμε τώρα. Ευχαριστώ. Έχετε ερωτήσεις για την μεταφορά πιστώσεων υπαριθμών 58. Όχι υπέρ κατά αποχές μία αποχή εγκρίνεται 61 Έχουμε την 60 λέει ο κύριος Σούργιαν η οποία είναι προβληματική μία νέα πρόταση για να αντιμετωπίσουμε τον πανανικό θέμα. Επειδή η καταγλυκτική προθεσμία είναι τον Ιανουάριο. Και δεν έχουμε ακόμα νομική φάση. Ίσως μπορούμε να αναβάλουμε αυτή την απόφαση παρόλα αυτά που ανέφερα προηγουμένως. και ίσως στον τριγωνικό διάλογο κύριε Πρόεδρε μπορείτε να θίξετε αυτό το θέμα για, τις νομική, για τη νομική βάση για το θέμα αυτό γιατί αυτό εναπόκειται στο Συμβούλιο. Αν έρθει η νομική βάση και μπορούμε να έχουμε μια συνεδρίαση της Επιτροπής μας την επόμενη εβδομάδα ή και αργότερα, εντάξει. Αλλιώς, ακόμα και αν εγκριθεί μεταφορά, τα χρήματα αυτά θα χαθούν. Γι' αυτό προτείνω να περιμένουμε και να δούμε. Ωραία, λέω. Αν συμφωνείτε να περάσω και στην επόμενη, Πρόεδρος, για την μπανάνα. Ε, αυτή η περιπέτεια της μπανάνας περιπλέκεται. Ίσως να ακούσουμε και την άποψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χάιντερ, θέλεις τον λόγο. Απλώς για να ζητήσω από την Κομισιόν να μας ε, εξηγήσει τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση. Αν δεν υπάρξει νομική βάση, τι θα γίνει. Γιατί οι διαπραγματεύσει κανονικά είναι μεταξύ Συμβουλίου και ημών. Πράγματι, αυτό ήθελα να ζητήσω και εγώ από την Κομισιόν. Είναι πολύ πολύπλοκα τα μπανανικά. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για το θέμα αυτό της νομικής βάσης. Μας είπαν ότι ήταν πάρα πολύ κατεπήγον να βρούμε πόρους για τον τομέα αυτό και είμαστε στο τέλος του έτους και δεν υπάρχει νομική βάση. Λοιπόν, ήταν σχετική και αυτή η έννοια του κατεπήγοντος από ό,τι φαίνεται. Θέλει να δώσει την άποψη της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Όντως, η πρόταση μεταφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν να βάλουμε στη νέα γραμμή για τα συνοδευτικά μέτρα υπέρ των μπανανοπαραγωγών στις χώρες ΑΚΕ ε, το ποσό αυτό, διότι από πού προέρχονται οι πιστώσεις που είναι να μεταφορθούν, ε, ε, μην ξεχ... εντάσσονται μάλλον σε μια συμφωνία που συνήθει στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής για τον διορθωτικό προϋπολογισμό υπαριθμών 3. Τελικά δεν συμφωνήσαμε για όλα τα υπόλοιπα και κατέπεσε και αυτό, οπότε δεν υπάρχει ουσιαστικά διορθωτικός προϋπολογισμός και προτείναμε εμείς να βάλουμε τα ποσά στη γραμμή της μπανάνας ελπίζοντας ότι η νομοθετική διαδικασία, δηλαδή ε, τα περί νομικής βάσεως, ε, θα ολοκληρώνονταν μέχρι το πέρας του τρέχοντος. Όμως, αν δεν συμφωνήσουμε για την νομική βάση, τι σημαίνει αυτό. Ακόμη και αν εγκρίνουμε την μεταφορά, η πίστοση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 2010. Άρα... Θα είναι άχρηστη η πίστοση. Ε, νομίζω ότι ο εισηγητής το ανέφερε, θα το αναφέρει αυτό στον τριμερή διάλογο την επόμενη εβδομάδα. Ε, νομίζω ότι είναι επικοδομητική αυτή η προσέγγιση γιατί έτσι θα δούμε σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε. Ε, να δούμε δηλαδή αν υπάρχουν δυνατότητες να ολοκληρωθεί τελικά ε, φέτος η νομοθετική διαδικασία και εν η αυτή περίπτωση μπορούμε να επανεξετάσουμε την πρόταση που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μεταφορά της πίστοσης. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Από την άποψη των ποσών, των ποσών αυτό αντιπροσωπεύει στις μεταφορές ένα εκατομμύριο. Όχι, πληρωμές, πληρωμές. Ένα μισή εκατομμύριο ευρώ. Ένα μισή εκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή, αν τα χρήματα αυτά δεν χρησιμοποιηθούν, θα επιστρέψουμε 1,5 εκατομμύριο παραπάνω στα κρατημέλη. Πράγμα Τι θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, ναι, θέλω να διευκρινίσω αυτό που είπατε για τις πιστώσεις πληρωμών, αλλά για τις πιστώσεις υποχρεώσεων πρόκειται σχεδόν για 70 εκατομμύρια. Και αυτά τα 70 εκατομμύρια αν δεν υπάρξουν το 2010 και τα μέτρα τα συνοδευτικά για την μπανάνα, θα πρέπει να τα βρούμε το 2011 και τα επόμενα χρόνια για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη συμφωνία που αφορά 190 εκατομμύρια για την περίοδο 2010-2013. Πράγμα το οποίο θα διεύρυνε τις δυσκολίες χρηματοδότησης των μέτρων αυτών. Γι' αυτό και υποβάλαμε αυτή την σε μεταφορές, γιατί αυτές οι πιστώσεις που υπάρχουν στον προπολογισμό 2010 του δίνουμε την ευκαιρία να χρησιμοποιηθούν. Και αν δεν χρησιμοποιηθούν, όπως είπατε, θα χαθούν. Και θα έχουμε πρόβλημα να εντοπίσουμε πού θα βρούμε 70 εκατομμύρια. Μια, μια, υπο, μια πίστοση δηλαδή υποχρέωση που είναι και η πραγματική δέσμευση. Ναι, είναι διόλο μελιτέο ποσό όσον αφορά τις πιστώσεις υποχρεώσεων. Εσείς είστε ικανοποιημένοι. Και, και ναι και όχι. Όχι γιατί δεν έχουμε ακόμα βρει μια λύση με την ε, νομική βάση. Αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και ενώπιον του κινδύνου να μην ξέρουμε τι θα γίνει με αυτό το ποσό γιατί δεν το βάζουμε το 1,5 εκατομμύριο στον τροποποιημένο προπολογισμό του ΕΤΑ. Ο εισηγητή θα μα πει ποια είναι τα δικά του συμπεράσματα, αλλά με μου φαίνεται ότι η πρόταση του εισηγητή να μην εγκρίνουμε σήμερα, γιατί δεν έχουμε νομική βάση, αλλά ενδεχομένω την επόμενη εβδομάδα μπορούμε να δούμε τι θα γίνει μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Αν έχουμε περισσότερε διευκρινήσει για τη δυνατότητα έγκριση μια νομική βάση, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία δήρηση επί της ουσίας για τη μεταφορά αυτή αν είναι απαραίτητη. Ο κύριος Σούριανο, η εισηγητής. Πρόεδρε. Ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα είναι σε θέση να διαχειριστεί αυτή τη νομική βάση, γιατί για μένα ως εισηγητή το 2010 δεν είναι κακό αν εξαφανιστούν όλα αυτά από τον προϋπολογισμό μου, αλλά Είμαι και μέλο τη Επιτροπή προπολογισμού και έχω να αντιμετωπίσω το πρόβλημα των συνόλων του προπολογισμού για το 2011. Αν αυτά τα 70 εκατομμύρια δεν τα βρούμε στο δικό μου προϋπολογισμό, απλώς όλα αυτά τα προβλήματα θα εμφανιστούν το 2011. Που είναι ούτως ή άλλως προβληματικός. Άρα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πιέσουμε το Συμβούλιο. Αυτή είναι η μόνη δυνατότητα. Όπως σας είπα, στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Προπολογισμού δεν θα είμαι παρόν, αλλά αν ο τριμερής διάλογος δώσει ένα θετικό μήνυμα, τότε ίσως θα ήταν λογικό να περιψηφίσουμε αυτήν την μεταφορά την επόμενη εβδομάδα. Να σας πω και για την επόμενη. Ναι, λοιπόν. Έτσι θα πράξουμε. Και όπως πρότεινε και η Κομισιόν, προτείνουμε να μπει στην ημερήσια διάταξη του τριμερούς διαλόγου της επόμενης Δευτέρας. Είμαι βέβαιος ότι ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα θέλει να βρει συμφωνία με το Συμβούλιο και γι' αυτό το σημείο με την ευκαιρία αυτού του τριγωνικού διαλόγου για τον οποίο, για τον οποίο δεν έχουμε και πολλή ουσία αλλά σιγά σιγά γεμίζουμε την ημερησία διάταξη. Συνεχίστε λοιπόν με το 61. Την 61. Στην 61 δεν έχω καμία παρατηρήση. Απλώς σας ζητώ να υπερψηφίσετε. Ωραία. Για την 61 λοιπόν, θέλει κανείς το λόγο, όχι. Ποιοι είναι υπέρ. Σας ευχαριστώ. Ποιοι είναι κατά. Δύο αποχές. Δεν υπάρχουν αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν και η 61. Voilà. Donc je comprends que nous avons d'autres euh, demandes de virement sur le budget. Έχουμε και άλλα αιτήματα μεταφοράς, αλλά που μπορούν να εξεταστούν κάπως αργότερα. Έχετε την ίδια άποψη. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, Πρόεδρε. 63 είναι τμήμα του μεγάλου πακέτου και δεν μπορεί να ψηφιστεί από μόνη της. Χωριστά. Μαζί είναι ο τροποποιητικό προπολογισμό 10 και η τροποποιητική επιστολή στον τροποποιητικό προπολογισμό 10 και ολόκληρο το πακέτο για του χρόνου. Αν ε, συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο και οριστικοποιηθείτε αυτή η συμφωνία. Φυσικά και θα το στηρίξω αυτό, αλλά όχι τώρα. Ωστόσο, για να επιταχύνουμε το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας, η 64 δεν έχει πρόβλημα, μπορεί να ψηφιστεί και τώρα. Και έχουμε και το Info 3 που μπορεί επίσης να ψηφιστεί. Αλλά και έχω μια παρατήρηση να κάνω. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, για τον εισηγητή λοιπόν η 64, η μεταφορά 64 μπορεί να ψηφιστεί σήμερα. Να σας ρωτήσω όμως, γιατί τη λάβαμε μόλις την Παρασκευή και δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να το, να το μελετήσετε. Έχετε αντίρρηση να ψηφίσουμε αυτή την τροπολογία, τη μεταφορά. Ωραία. Ψηφίζουμε και για την 64 τότε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Μία αποχή. Η 64 λοιπόν εγκρίνεται. Άλλο. Λάσλο. Ναι. Έχουμε αυτό το info 3. το υποστηρίζω εγώ, αλλά πρέπει να κάνω μια παρατήρηση, ότι είναι μια μεταφορά από το τουρκοκυπριακό πρόγραμμα. Και εγώ μιλώ στο όνομα του δικό μου ως αλλά ξέρω και την άποψη του κύριου Μπέγκε, που ενδιαφέρεται πολύ για τα τουρκοκυπριακά ζητήματα. Και είναι επίσης έτοιμος να το δεχτεί, αλλά με την εξής παρατήρηση. Εάν ένα πρόγραμμα στο τουρκο-κυπριακό θέμα είναι, έχει μπλοκαριστεί και δεν υπάρχει τρόπος να δαπανηθούν τα χρήματα, υπάρχουν άλλα προγράμματα στο ίδιο πλαίσιο. Γιατί να μην δοθούν τα χρήματα εκεί και όχι σε ένα τελείως διαφορετικό ζήτημα. Είναι μια συμβουλή δηλαδή για το μέλλον ή ένα αίτημα από τη δική μας πλευρά ότι αν ε, τρέχουν διάφορα προγράμματα παράλληλα, αυτό που μπλοκάρεται να μην δαπανώνται τα χρήματα σε τελείως διαφορετικό τομέα, αλλά να δαπανώνται σε κάποιο παραπλήσιο πρόγραμμα, γιατί διαφορετικά οι στόχοι του προπολογισμού δεν πληρούνται αν είναι αυτό δυνατό. Αλλά και πάλι πρόκειται για μια γενική φύση παρατήρηση. Μπορούμε να ψηφίσουμε ωστόσο για την πρόταση. Ε, ναι. Να θυμίσω πως αυτή η μεταφορά έχει ως αντικείμενο να πάρει χρήματα πιστώσεις πληρωμών από ένα κεφάλαιο βοήθειας προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα 1.910.000 ευρώ γιατί αυτά τα χρήματα δεν μπορούν να δαπανηθούν υπέρ του προγράμματος που είχε προβλεφθεί φέτος έτσι ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για διάφορα κεφάλαια ε, ενημέρωσης και πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κυρία Βέρμαν και ο κύριος Χαρτόγκ έχουν ζητήσει το λόγο. Θέλω να κάνω μια σύντομη παρατήρηση. Μίλησα προηγουμένως με κάποιο εκπρόσωπο της Κομισιόν. Δεν θα χαθούν τα χρήματα για την τουρκικο-κυπριωτική ε, κοινότητα. Απλώς δεν μπορούν να δαπανηθούν τώρα και όταν τελειώσει αυτό το πρόγραμμα νομίζω ότι θα, λάβουν, θα λάβει η τουρκοκυπριακή κοινότητα τα χρήματα. Αυτό κατάλαβα από, την, ε, τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Αυτό ήθελα να σας αναφέρω σε όλους. Σας ευχαριστώ. Επομένως υποστηρίζετε <clears throat> αυτή τη μεταφορά εσείς η ίδια. Μπορώ να δεχτώ ότι όπως έχουν τα πράγματα τώρα, τα χρήματα θα δαπανηθούν με διαφορετικό τρόπο. Δεν υποστηρίζω απόλυτα τον τρόπο με τον οποίο θα δαπανηθούν πάντως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτή την ε, ε, διευκρίνηση. Κύριο Σαρτόμπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να θέσω και ένα σύντομο ερώτημα προς την Κομισιόν. Θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά για επικοινωνία και πληροφόρηση σε σχέση με τη μελλοντική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς. Και δεύτερη ερώτηση. Πώς συνδέονται όλα αυτά με τη μελλοντική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Δούναβη με το ποδήλατο. Ναι, ναι, αυτό είναι το, το σχέδιο, λέει ο, <clears throat> ο Λαμασούρ. Ενδιαφέρον, ενδιαφέρον. Μπορεί να μα διαφωτίσει η Κομισιόν για τον ποδηλατικό γύρο του Δούναβη. Ευχαριστώ. Πράγματι, η μεταφορά ποσών είναι πράγματι για να ενισχυθεί η επικοινωνία και η πληροφόρηση και να αντιμετωπιστούν ανάγκες οι οποίες ε, ανέκυψαν περισσότερο από αυτό το οποίο προβλεπόταν. Ο στόχος είναι να γίνει πιο γνωστή η Ευρωπαϊκή Ένωση στις υποψήφιες χώρες και να ευαισθητοποιήσουμε τον πληθυσμό σε σχέση με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το Δούναβι με ποδήλατο μπορώ να σας στείλω ένα σύνολο, ε, σε σύνοψη το σύνολο των δραστηριοτήτων οι οποίες ε, προβλέπονται. Κατά τα άλλα δεν έχω στοιχεία να σας δώσω αυτή τη στιγμή, αλλά μπορώ να σας ε, στείλω εγγράφως μια περιγραφή όλων αυτών των δραστηριοτήτων. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Από ό,τι θυμάμαι, αυτό το πρόγραμμα Δούναβης με το ποδήλατο προέρχεται από μια τροπολογία του Κοινοβουλίου. Θα μας δώσετε εσείς όμως τις λεπτομέρειες για τις συγκεκριμένες δράσεις που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια του προγράμματος. Είναι υπέρο η ηγητή. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ για την ε, μεταφορά. Υπέρ. Κάτα. Αποχές. Μία. Ποιος βέρτε μας. Απέχει. Ευχαριστούμε. Λάσλο Σούριαν. Ο Λάσλο Σούριαν εκπλήρωσε την αποστολή του και τώρα θα στραφώ στον ε, Βλάντιμιρ Μάνκε και εκείνο έχει να μας προτείνει κάποιες μεταφορές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχουν ε, δέκα μεταφορές για τα λοιπά τμήματα. Ε, μία μόνο όμως χρειάζεται να σας εξηγήσω γιατί οι άλλες είναι παρεμφερείς. Ε, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή μεταφορά 7, το δικαστήριο όπως και τα λοιπά θεσμικά όργανα πρέπει να αντισταθμίσει ε, τους μη καταβληθέντες ε, μισθούς. Το θυμάστε ε, το, την αύξηση του 1,85% που πρότεινε η Επιτροπή και απέριψε το Συμβούλιο και τελικά κατατέθη αγωγή ενώπιον του δικαστηρίου για κύρωση της απόφασης. Ε, στις 24 Νοεμβρίου το δικαστήριο ακύρωσε τελικά την απόφαση του Συμβουλίου και γι' αυτό πρέπει να εγκρίνουμε αυτήν την μεταφορά καθώς και όλες τις υπόλοιπες που εντάσσονται ε, σε αυτόν τον τομέα. Πρόεδρε, υποθέτω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, θα ε, ακολουθήσει, θα συμμορφωθεί μάλλον με την απόφαση του δικαστηρίου και θα ζητήσει την εφαρμογή της αύξησης του 1,85, ε, δηλαδή 6,8 εκατομμύρια, εκ των οποίων 0,8% είναι οι μη καταφυγέντες μισθοί μέχρι το, τον Ιούνιο του 2010 Ε, και αντίστοιχο ποσό για το 2009 ε, πάλι για τους μισθούς. Οπότε ζητώ να ε, εγκρίνετε αυτή τη μεταφορά. Ευχαριστούμε. Συγγνώμη, μιλάμε για τις δύο αποφάσεις του δικαστηρίου. θα σας εξηγήσω την επόμενη. Ας ψηφίσουμε ίσως πρώτα για αυτή τη μεταφορά. Ωραία. Ο κύριος Αρτόν έχει ζητήσει το λόγο. Πρόεδρε, λέγεται ότι η νομική υπηρεσία του Δικαστηρίου της Ένωσης θα πρέπει να ζητήσει και άλλες νομικές γνωμοδοτήσεις, κάτι που δεν έγινε την εποχή που προετοιμάζαμε τον προϋπολογισμό. Ε, δηλαδή θα, ζητή, θα ζητηθούν εξωτερικές εγγνωμοδοτήσεις. Σε, τι, γιατί ακριβώς γίνεται αυτό. Ε, la Cour de Εκπροσωπείτε μήπως το δικαστήριο. Α, ο κύριος Σιμονέτη, παρακαλώ. Σα Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την μεταφορά πιστώσεων υπαριθμών 7 όπως εξήγησε και ο εισηγητής σας Πρόκειται για το 1,85% την αύξηση αυτή των μισθών που βέβαια δεν προβλεπόταν στον προϋπολογισμό του 2010. Προτείνουμε, χάρη σε διάφορες εξοικονομήσεις που έχουμε στον αντίστοιχο τίτλο αλλά και επί τη βάση προβλέψεων που υπήρχαν στον προπολογισμό για την αύξηση των μισθών από τον Ιούλιο του 2009, προτείνουμε να συλλέξουμε τα απαραίτητα κονδύλια για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την αναπροσαρμογή των ε, μισθών εφόσον αποφασίσει το Συμβούλιο ενδιαμέσως. Υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία ήταν αβέβαια όταν κάναμε αυτή την πρόβλεψη. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που απέριψε τη θέση του Συμβουλίου όπως είναι γνωστό και το δεύτερο στοιχείο αβεβαιότητας είναι η απόφαση του Συμβουλίου το οποίο πρέπει <clears throat> να εγκρίνει αυτή την ε, αναπροσαρμογή των ε, μισθών. Εάν γίνει δηλαδή, λοιπόν αυτή η απόφαση, θα πρέπει να βρίσκονται στην αρμόδια γραμμή του προπολογισμού για να μπορούν να καταβληθούν τα χρήματα αυτά. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η μεταφορά και για το ε, δικαστήριο και για, άλλους, ε, για άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει όλοι να είναι έτοιμοι να καταβάλουν τα ποσά αυτά. Ε, από τη στιγμή που το Συμβούλιο θα πάρει την αρμόδια απόφαση. Ευχαριστώ. Ναι, ναι. Ένα λεπτάκι. Θα σας δώσω το λόγο κύριε Άρτον. Το δικαστήριο εφίσταται τη συνέπειες ουσιαστικά της δικής του απόφασης. Αυτό, αυτό μας εξηγήσατε μόλις. Κάθε όργανο τι προσπαθεί να κάνει τα λεφτά που περισσεύουν ε, στα τέλη του 2010 και διακόπτει ο πρόεδρος μάλιστα κατάλαβα καλά και επανέρχομαι στον κύριο Άρτον. Δεν απαντήσατε στην ερώτησή του ρώτησε για την αύξηση ή μάλλον ρωτήσατε γιατί το δικαστήριο πλέον ε, ζητά εξωτερικές ε, γνωμοδοτήσεις. Δεν, δεν έφερε επί της μεταφοράς η ερώτηση του κ. Αρτών. Απάντηση. Νομίζω υπάρχει παρερμηνία ε, ο συνάδελφος από το ελεγκτικό συνέδριο που είναι δίπλα μου μου λέει ότι εκείνοι έχουν ε, ε, θέσει τέτοιο θέμα. Το δικαστήριο δεν μας αφορά δηλαδή αυτό το θέμα. Θα απαντήσει ο συνάδελφος. Εκτός μικροφώνου ο Πρόεδρος. Oui. Nous allons revenir à la question. Θα επανέλθουμε στην ερώτηση του κ. Άρτον για το ελεγκτικό συνέδριο. Για το δικαστήριο μας διαφωτίσατε. Είναι υπέρ ο εισηγητής. Ψηφίζουμε. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Ευχαριστώ. Οπότε η μεταφορά 07 του δικαστηρίου εγκρίνεται. Τώρα ας περάσουμε στην 8. pán eh, eh, Ευχαριστώ. Αν συμμορφωθεί με την απόφαση του δικαστηρίου το Συμβούλιο, θα καταπέσει η 8. Ε, σε τι αναφέρεται αυτή η μεταφορά ποσά που ε, υπολείπονται ε, σε διάφορες γραμμές του προϋπολογισμού. Εάν δεν ε, εκταμιευθούν, τότε το δικαστήριο θα χρησιμοποιήσει αυτά τα ποσά για να ε, πληρώσει την εκμίσθωση του κτηρίου του. Ε, θα πρότεινα να υπερψηφίσουμε αυτό το αίτημα μεταφοράς υπό την αίρεση βεβαίω ότι το Συμβούλιο δεν θα συμμορφωθεί με την απόφαση του δικαστηρίου. Άλλη εναλλακτική λύση είναι να μην ναι, ψηφίσουμε σήμερα και να περιμένουμε να εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου και να επανέλθουμε στο τέλος του 2010 ε, σε αυτό το θέμα. Εγώ προτιμώ τη δεύτερη εναλλακτική λύση που προτείνατε. Μου φαίνεται πιο λογική. προσωπική μου άποψη. Ε, είναι, αλλιώς θα φάσκουμε και αντιφάσκουμε με αυτές τις δύο πιστώσεις. Έχουμε υπερψηφίσει ήδη την μεταφορά 7, πολύ ωραία, και προτείνει το δικαστήριο με φυή τρόπο να χρησιμοποιήσει αυτό το περιθώριο λιγμών που έχει και αν δεν ευοδοθούν οι προσπάθειες τότε να ασχοληθούμε και με την 8. Αυτά για το δικαστήριο. Τώρα, ε, Πάμε στο ελεγκτικό συνέδριο. Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ε, εξετάσουμε από κοινού όλες αυτές τις μεταφορές που βασίζονται στην απόφαση του ΔΕΚ. Δηλαδή έχουμε ε, τρεις ε, μεταφορές για την ΟΚΕ ε, δύο, μάλλον τρεις για το ελεκτικό συνέδριο. Μετά έχουμε την Επιτροπή των Περιφερειών, V5 ε, 2010. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, C12, μπορεί να μην το έχετε στο φακελό σας, αλλά είναι στην ίδια κατηγορία. Όλες αυτές οι μεταφορές είναι μία ή ίδια κατηγορία μεταφορών και προτείνω να τις ψηφίσουμε όλες από κοινό. Υπάρχει μόνο το θέμα των ε, μεταφορές C12 του Κοινοβουλίου γιατί οι γραμμές όπως το κεφάλαιο 13 συνεδριάσεις και διασκέψεις από όπου πρέπει να προέλθουν αυτά τα χρήματα έχει χαμηλό ποσοστό απορρόφησης λόγω της αλλαγής στον κανονισμό. Όταν άλλαξε ο κανονισμός είχαμε μια διευθυντική αλλαγή και άρα το ερώτημά μου είναι τι θα συμβεί στο 2011. Θα υπάρξει μείωση των ποσών στο, 13, στο κεφάλαιο 13. Δεν ξέρω αν έχει γίνει ήδη αυτή η μείωση για το 2011. Και βεβαίως είμαι υπέρ όλων αυτών των μεταφορών που είναι παρόμοιες. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Πριν να ψηφίσουμε λοιπόν τώρα για αυτές τις μεταφορές, να επανέλθω στο θέμα του κυρίου Χάρτονγκ στην ερώτησή του. Δηλαδή, η ερώτηση που έκανε ο κύριος Χάρτονγκ περισσότερο αφορούσε το ελεγκτικό συνέδριο παρά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εγώ δεν κατάλαβα καλά και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι έτοιμο να απαντήσει. Του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά την, ε, το αίτημα μεταφοράς ε, υπαριθμών 7, όπου θέλουμε πιστώσεις για νομικούς συμβούλους. Έχουμε ένα μικρό ποσό στον προπολογισμό μας, 20.000 ευρώ ετησίως, για εξωτερικές νομικές ε, συμβουλές. Κατά τη διάρκεια του 2010 χρειαστήκαμε Είχαμε περισσότερες υποθέσεις από ό,τι στο παρελθόν και γι' αυτό χρειάζεται να προσθέσουμε ακόμα 16.000 σε αυτό το ποσό. Οι νομικοί σύμβουλοι χρησιμοποιούνται είτε για επίλυση θεμάτων ελέγχου, δηλαδή για, ας πούμε για εταιρείε οι οποίες ε, δεν μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν σωστά τα χρήματα της Ένωσης, ε, που θα πρέπει να, να ονομάζονται στις εκθέσεις ε, των ε, του, του ελεγκτικού συνεδρίου. Σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε ε, νομικές συμβουλές από νομικούς που αφορούν διοικητικά ζητήματα. Τώρα, η αύξηση του κόστους είναι διοικητικό ζήτημα και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι χρησιμοποιούνται οι συμβουλές αυτές για να προστατεύσουμε τα οικονομικά συμφέροντα της κοινότητας σε μια περίπτωση η οποία, με την οποία ασχολούμεθα. Μάλιστα, ευχαριστώ. Ε, si vous permettez une remarque euh, αν μου επιτρέπετε μια παρατήρηση από τη δική μου προσωπική ιστορία για το ελεγκτικό συνέδριο και το λέω για τον κύριο Αρτών και το ελεγκτικό συνέδριο. Εγώ ξεκίνησα την επαγγελματική μου σταδιοδρομία ως υπάλληλο εισαγγελέα στο γαλλικό ελεγκτικό συνέδριο πριν από μισό αιώνα. Τότε λοιπόν, για να κρίνει κανείς την ποιότητα ενός εισαγγελέα, μας πλήρωναν με πριμ, ανάλογα με την απόδοσή μας. Ποια ήταν η απόδοση. Τα ποσά που ξαναφέρναμε στον προπολογισμό του κράτους και τα οποία είχαν πέσει θύματα διασπάθησης. Άρα λοιπόν τα πρίμα αυτά τα έπαιρνε ο εισαγγελέα επιπλέον του ετησίου μισθού του. Και το λέω λοιπόν αυτό εδώ προς το ελεγκτικό συνέδριο και ίσως και ο κύριος Χαρτόγκο και άλλοι συνάδελφοι να θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα κριτήρια στο μέλλον. Μπορούμε να κρίνουμε την σωστή χρήση των επιπλέον κονδυλίων που ζητά το ελεγκτικό συνέδριο μετρώντας πόσα χρήματα ξαναβάζει στον ευρωπαϊκό προπολογισμό και πόσο περιορίζει τις πατάλες που σχετίζονται με αυτό εδώ το επιπλέον ποσό. Σας δίνω αυτή την προσωπική μου βήρα λοιπόν και αυτή την πρόταση. Ο κύριος Άρτον θέλει να πάρει και πάλι το λόγο ή όχι. Ναι, το είχατε ζητήσει, ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω εμείς ε, υποστηρίζουμε ιδιαίτερα την άποψη του ελεκτικού συνεδρίου και είμαστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τα χρήματα του φορολογούμενου. Γι' αυτό θέτω το ερώτημα αν χρειάζεται να έχουμε τόσες πολλές ε, διαδικασίες. Ωραία, λέει ο πρόεδρος. Πολύ καλή ερώτηση. Μπορούμε λοιπόν να θέσουμε όλες αυτές τις ε, μεταφορές σε ψηφοφορία από κοινού, κύριε Σιγητά, συμφωνείτε. για να είμαστε σίγουροι κύριε Σιγητά ότι δεν κάνουμε σφάλματα γιατί υπάρχουν πολλά θεσμικά όργανα και πολλές μεταφορές. Μπορείτε να μας υπενθυμίσετε ποιο είναι ο κατάλογος των μεταφορών που μπορούμε να ψηφίσουμε από κοινού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επαναλαμβάνω. Το ένα το κάναμε ήδη για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η 5 2010, δύο μεταφορές για το Ελεκτικό Συνέδριο, 05 και 06 για το Ελεκτικό Συνέδριο, Επιτροπή Περιφερειών, 5 2010, και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο C12. Όλα μαζί μπορούμε να τα ψηφίσουμε αυτά γιατί είναι ταυτόσιμες οι μεταφορές και νομίζω ότι όλοι θα ψηφίσουν με τον ίδιο τρόπο. Ωραία. Ψήφι υπέρ αυτών των μεταφορών. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται λοιπόν οι μεταφορές αυτές. Μένουν μερικές ακόμα κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να απαντήσει το ερώτημά μου. Θα το ξαναθέσω <clears throat> για τη μεταφορά C12 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όλα τα θεσμικά όργανα έχουν εξοικονομήσει χρήματα για να καλύψουν αυτές τις μεταφορές. Αυτό που έχει κάνει όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ότι έχει αλλάξει ορισμένου κανόνες και χάρη σε αυτούς έχει υπάρξει μια εξοικονόμηση. Θα ήθελα να ξέρω αν αυτοί οι νέοι κανόνες έχουν ληφθεί υπόψη αλλιώς θα έχουμε πάλι πρόσθετα χρήματα το 2011. Ναι, ναι. Ψηφίσαμε το... τη μεταφορά, αλλά θέλει να θέσει ένα ερώτημα ο κύριος Συγητής για το 2011. Κύριε Πρόεδρε, πράγματι η αλλαγή των κανόνων οδήγησε σε εξοικονομήσεις. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Προηγουμένως δεν είχαμε κάποια τέτοια ενέργεια για τον προϋπολογισμό του 2011. Βασιστήκαμε ήδη στην κεκτημένη εμπειρία και έλαβαν υπόψη αυτή την τροποποίηση των κανόνων για να μπορούμε να έχουμε προβλέψεις οι οποίες είναι πιο σύμμορφες με την πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την απορρόφηση των κονδυλίων. Σας επιβεβαιώνω λοιπόν για το 2011 έχουμε λάβει υπόψη αυτή την τροποποίηση. Πολύ ωραία λέει ο πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σιγητά, άλλες ε, μεταφορές. <clears throat> ναι, θέλω να ευχαριστήσω τον ε, εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου για τα θέματα αυτά. Και τώρα κύριε Πρόεδρε, θέλω να έρθω στη μεταφορά του κυρίου, του κυρίου Χάρτοκ, VAV 07 του Ελεκτικού Συνεδρίου. Νομικά έξοδα. <clears throat> Εξωτερικές νομικές εμπειρογνωμοσύνης. Ήταν περισσότερε από ό,τι προβλεπόταν, γι' αυτό γίνεται αυτή η αίτηση και αυτή η εξήγηση που θέλω να δώσω στον κύριο Χάρτον. Υποστηρίζω την ε, μεταφορά αυτή. Πολύ ωραία, λέει ο πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Ακούσαμε λοιπόν και την απάντηση του ελεκτικού συνεδρίου. Ψήφι υπέρ της V07. Ε, Κατά. V07 07 ψηφίζουμε. Ευχαριστώ. Αποχές. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται λοιπόν η μεταφορά αυτή. Κύριε Σιγητά, συνεχίζουμε. Έχουμε την 32010 τη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. 15.000. Γιατί είχαν πάλι μεγαλύτερα, μεγαλύτερο κόστος ε, σε νομικό επίπεδο. Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς ε, αλλά έχω και ένα ερώτημα προς την Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή. Λένε ότι 80% όλων των πόρων τους στον τομέα αυτό δαπανήθηκαν σε μια έκτακτη περίπτωση. Μπορείτε, μπορεί να μας πούν τι ήταν αυτή η νομική περίπτωση στην οποία δαπανήσαν τα λεφτά αυτά ήτανε. Μπορεί ο εκπρόσωπος της ΟΚΕ να απαντήσει. Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω. Θα πρέπει να το συζητήσω με την νομική μας υπηρεσία. Όπως είπαμε όμως, οι αρχικές πιστώσεις ήταν 40.000 ευρώ, 32.000 ήταν το 80% αυτού, δηλαδή ακόμα και σε μια νομική διαδικασία δεν είναι τεράστιο ποσό η δυσκολία με αυτό το άρθρο είναι ότι σε φυσιολογικά έτη δεν ε, χρησιμοποιούμε τις πλήρες πιστώσεις και για να μην έχουμε ποσά τα οποία μένουν αδαπάνητα κάνουμε αιτήσει οι οποίες αφορούν το μέσο κόστος των δικαστικών διαδικασιών αλλά εφέτος το ξεπεράσαμε το αρχικό αυτό ποσό και γι' αυτό κάνουμε την αίτηση για τη μεταφορά αυτή για να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε το πρόσθετο κόστος. Σας ευχαριστώ. Θεωρείτε κύριε Σιγητά ότι μπορούν να, να προχωρήσουμε με αυτή την ε, απάντηση χρειάζεται πιο πολύ χρόνο γιατί θα συνεδριάσουμε και την επόμενη εβδομάδα. Πρόεδρε. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να υπερψηφίσουμε σήμερα τη μεταφορά. Θα ήθελα όμως ε, να απαντήσουν γραπτός. Να μας απαντήσουν γραπτός από την ΟΚΕ. Τι έγινε με αυτό το 80% των ε, πιστώσεων. Ε, σε τι δαπανήθηκαν. Très Ποιοι είναι υπέρ της μεταφοράς 3. Κατά. Αποχές. Καμία. Εγκρίνεται. Ε, πάλι για την ΟΚΕ. Έχουμε τη μεταφορά 4. Μάλιστα. Πρόεδρε, ε, η μεταφορά αυτή συνδέεται με τη μεταφορά της 9ης Δεκεμβρίου που υπερψηφίσαμε για την Επιτροπή των Περιφερειών. Ε, σχετίζεται με έναν έλεγχο ε, ασφαλείας Ε, για να αντικαταστήσουμε τον απαρχαιωμένο ε, εξοπλισμό ε, με νέο εξοπλισμό. Μάλιστα, δεν υπάρχει καμία ερώτηση. Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ, για τη μεταφορά 4, για την ΟΚΕ. Ευχαριστώ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έχετε και άλλες μεταφορές κύριε Σιγητά. Áno, ešte δύο για το ε, τελευταία στιγμή βέβαια μεταφορές ε, αγορά ενός κτηρίου στη Σόφια, είναι η μία μεταφορά και σχετίζεται με την έκθεση της κυρίας Χολμάιερ προτείνω να αναβληθεί για τις 8 Δεκεμβρίου όταν εξετάσουμε και την έκθεση της κυρίας Χολμάγερ. Αναβολή κατά μία εβδομάδα λοιπόν και τέλος η 14 και πάλι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Προεδρείο ενέκρινε μία μεσοπρόθεσμη στρατηγική για την ε, πληροφορική και τους σχετικούς εξοπλισμούς και το πρόγραμμα αυτό συνάδει με την στρατηγική αυτή. Εάν εγκρίνουμε αυτή την μεταφορά θα εξοικονομήσουμε χρήματα για το 2011. Καλύπτονται τέσσερα προγράμματα με τη μεταφορά ε, ο εξοπλισμός για τις ψηφοφορίες στο Στρασβούργο που ε, είναι απαρχαιωμένος και πρέπει να αντικατασταθεί. Ε, τα, επιτοπλίστων ε, χρειάζεται να αντικαταστήσουμε μάλλον ε, σχεδόν όλο τον εξοπλισμό για τις ψηφοφορίες γιατί δεν λειτουργεί πια καλά κατόπιν ε, να αυξήσουμε την δυνατότητα χωρητικότητας αποθήκευσης βιντεοαρχείων Ξαναλέω ότι όλα αυτά εντάσσονται στη μεσοπρόθεσμη στρατηγική για την ε, τεχνολογία της ε, πληροφορικής και τα κονδύλια αυτά έχουν ήδη συμπεριληφθεί για το 2011. Οπότε, ε, ρωτώ, αν εγκρίνουμε σήμερα τις μεταφορές, θα ενταχθούν τα κονδύλια στις γραμμές του προϋπολογισμού του 2011. Très bien, je comprends. Donc, il y a une... Υπάρχει λοιπόν αυτό το ερώτημα, σας δίνω το λόγο. <clears throat> Απλώς αυτό το οποίο κατάλαβα είναι ότι ο εισηγητής μας προτείνει να αναβάλουμε την εξέταση του σε 13 που έχει να κάνει με την κτηριακή πολιτική και φυσικά και με την έκθεση της κυρίας Ολμαγέρ. κυρία Ολμαγέρ μου ζήτησε συγγνώμη διότι για λόγους ε, μεταφορών και δυσκολιών συγκοινωνιών δεν μπορεί να φτάσει ως το τέλος της συνεδριασής μας. Θα επανέλθουμε λοιπόν στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδριασής μας μαζί με το ΣΕ 13. Για το 14 το ίστατο και λουκούμιο λοιπόν θέμα θέτω αυτό το ερώτημα στις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ μόνο για μία διευκρίνηση. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξετάζουμε τον προϋπολογισμό του 2012. Τα τις προβλέψεις. Οι δαπάνες αυτές προβλεπόντουσαν για το πρώτο εξάμεινο του 2012. Σας επιβεβαιώνω ότι υπάρχει μια εξοικονόμηση η οποία θα εμφανιστεί μόνο το πρώτο εξάμεινο του 2012. 12 όχι 11. Θα έχουμε 10 εκατομμύρια λιγότερα στον προπολογισμό του 2012 εάν χρηματοδοτήσουμε από τα υπολείμματα του 2010 αυτή την ενέργεια. Κάτι σαν και αυτό που έκανε η Κομισιό με το ΙΤΕΡ δηλαδή. Χρειάζομαι να δαπανίσω το 2012, οπότε χρησιμοποιώ τα ρέστα μου από το 2010 για να τα καλύψω τα ποσά αυτά. Λοιπόν, τώρα τα απλοποιώ λιγάκι, όχι με, δεν σας τα λέω επιστημονικά όλα αυτά. Μετά από αυτή τη, τη διευκρίνηση, κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ. Ναι. Το καταλαβαίνω. Αλλά αυτό που κάνουμε είναι εμπροστοφόρτωση, προκαταβολή, προχρηματοδότηση. Κάνουμε μια επένδυση η οποία θα μας οδηγήσει σε μια... Α, κανονικά θα πρέπει να οδηγήσει σε εξοικονομήσεις του χρόνου. Γιατί το κάνουμε εφόσον πρόκειται για το 2012. Ό,τι κάνουμε φέτος πρέπει να δοκιμήσει του χρόνου. Γιατί το 2012. Ευχαριστώ. Κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μην αφήνει για αύριο αυτό που μπορεί να κάνει σήμερα, λέμε εμεί στην Πορτογαλία. Και στην Ελλάδα εξάλλου. Και νομίζω ε, ε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λαϊκή ρίση και εδώ. Πρέπει να εκπληρώσουμε τους στόχους του Κοινοβουλίου. Είναι κανόνας καλής διαχείρισης, χρηστής διαχείρισης να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα που έχουμε, ούτω ώστε να μην υπερφορτώσουμε του επόμενου προπολογισμού, Εφόσον έχουμε αυτή την ανάγκη, ελοχεύει ο κίνδυνο να υπάρχουν προβλήματα αφού να υπάρχει εξοπλισμός για τις ψηφοφορίες. Εμείς θεωρούμε ότι εφόσον έχουμε διαθέσιμα κονδύλια πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Τώρα αν γίνουν περικοπές στον προϋπολογισμό το 2011 ή και το 2012... Είναι ένα θέμα που μας ανησυχεί. Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να ανακουφίσουμε, να μην υπερφορτώσουμε τους επόμενους προϋπολογισμούς αφού τα έχουμε τα κονδύλια. Υποστηρίζουμε λοιπόν αυτό το αίτημα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος ε, Χάρτον έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, χαίρομαι που αναβάλαμε τη C13 για την επόμενη εβδομάδα. Για το C14 αυτό το κτίριο στη Σόφια θα κοστίσει 10 εκατομμύρια και θα έχουμε και 13 εκατομμύρια ε, για την ανανέωση του εξοπλισμού πληροφορικής. Αλλά, συγγνώμη, δεν είναι, προσ... Ε, ε, δεν είναι κόλαφος για τις οικογένειες στην Ιρλανδία. Ας είμαι λιγότερο κινητικός στις Βρυξέλλες, αν μπορούμε να βοηθήσουμε μια οικογένεια που απειλείται με έξωση στην Ιρλανδία. Τώρα πώς τα συνδέσατε αυτά τα δύο δεν είναι προφανή η σύνδεση ανάμεσα στα δύο σημεία. Τι λέει ο εισηγητής. Ε, αναβάλαμε τη C13. Θα σχολιάσω μόνο τη C14. Ε, η πρόθεσή μας για σήμερα είναι να ε, εγγραφεί αυτό στον προπολογισμό το 2012 γιατί για τότε έχει προβλεφθεί η επένδυση αυτή ε, την ανα, τις ανακαινήσεις ούτως ή άλλως δεν θα τις κάναμε το 2011. Εγώ είχα καταλάβει τουλάχιστον ότι προβλέπονταν όλα αυτά για το 2012. Ε, και εφόσον δεν έχουμε... Δεν, έχουμε, δεν υπάρχει αντικείμενο ουσιαστικά για να κάνουμε αυτές τις δαπάνες ε, γι' αυτό προτείναμε τη μεταφορά. Ε, θα το είχαμε προγραμματίσει για το 2011, μα ήταν για το 2011, έτσι δεν είναι. Ε, πρόεδρε, δεν έχω πρόβλημα ε, να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πιστώσεις τώρα αλλά ε, θέλω να ξέρω αν έχει προβλεφθεί η επένδυση για το 2011. Ποια ήταν η αρχική πρόθεση. Όταν ε, ε καταρτήσαμε τον προπολογισμό του 2011 δεν είχαμε πει ότι θα γινόταν η επένδυση το 2012 και πάλι ο κύριος Φερνάντες τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ίσως η Γενική Διεύθυνση για, τα, για τον πληροφορικό εξοπλισμό θα πρέπει να μας απαντήσει αλλά μπορούμε ήδη να ξεκινήσουμε από τώρα. Επομένως κερδίζουμε χρόνο και είμαστε πιο αποτελεσματικοί σε σχέση με τη χρησιμοποίηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού. Φαντάζομαι ότι μπορεί να προχωρήσει τώρα ήδη αυτή η επένδυση Ίσως όμως εδώ θα μπορούσε να μας τα διευκρινίσει τα θέματα αυτά η Γενική Διεύθυνση για τον πληροφορικό εξοπλισμό του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Ίσως ο, εγώ σας περιέπλεξα ένα πρόβλημα το οποίο είναι κάπως απλό. Είναι πιο απλό από ότι ένοχος είμαι αλλά έχω την επιστολή του Προέδρου Μπούζεκ. Και στην επιστολή αυτή εξηγεί ο κύριος Μπούζεκ, ο πρόεδρος Μπούζεκ, ότι αν χρησιμοποιήσουμε τώρα τα κονδύλια αυτά, θα επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να χρηματοδοτήσει αμέσως δαπάνες σε επίπεδο τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής και έτσι θα ελαφρώσει τον προϋπολογισμό του 2012 που μπορεί <clears throat> να αφιερωθεί σε άλλα θέματα. Αυτό θα λέγατε κύριε Λαφορέ, δεν είναι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε δύο στοιχεία στον προϋπολογισμό. Από τη μια μεριά υπάρχει μια βελτίωση των, των προϊόντων και από την άλλη πλευρά έχουμε συστήματα τα οποία είναι απειρχαιωμένα, τα οποία πρέπει να αντικατασταθούν όπως το σύστημα ψηφοφοριών και κάπως προκαταλαμβάνουμε μια επένδυση του 2012 και <clears throat> συνυπολογίζουμε την αύξηση ζήτησης για το 2012. Επομένως, ήδη κάνουμε κάποιες αγορές εξοπλισμού ώστε το 2010 και να μην χρειαστεί να γίνει το 2012. Γι' αυτό ήταν ατυχές αυτό που σας είπα προηγουμένως δεν βάσουμε χρήματα στο ψυχείο για να τα χρησιμοποιήσουμε το 2012, απλώς προκαταλαμβάνουμε εργασίες οι οποίες θα γινόντουσαν ούτως ή άλλως. Εντάξει, νομίζω ότι κατάλαβα και σας ζητώ συγγνώμη. Ω πρόεδρος πρέπει να κάνει σαφέστατα τα πράγματα και όχι να τα μπερδεύει. Ο κύριος Σαρτόκ και μετά ο συγητής θα μας πει τι θα κάνουμε. Κύριε Αρτόκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε το σύστημα ψηφοφορή, ηλεκτρονικής ψηφοφορίας λέτε ότι είναι απερχιαμένο. Εγώ βλέπω να δουλεύει μια χαρά. Πρέπει να σας πω ότι δεν πρέπει να κάνουμε δαπάνηση για πράγματα τα οποία δεν είναι απαραίτητο να αλλάχθουν. Είτε το 2011 είτε το 2012. Θα πρέπει να εξοικονομήσουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Σεγητά, ποια είναι η δική σας πρόταση. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι πρέπει να υπερψηφίσουμε αυτή τη μεταφορά. Αλλά... Θέλω να πω στον εκπρόσωπο της διοίκησης του Κοινοβουλίου Αν έχετε σχέδια για το έτος 1, 2, 3, 4, 5, δεν νομίζω ότι έχει νόημα να θέτε προτεραιότητα το 5 πριν από το 1. Είναι θέμα στοχοθεσία. Από τη στιγμή που έχουμε τι προτεραιότητε, θα πρέπει να τι διεξέλθουμε μία προς μία και όχι να τα κάνουμε ανάποδα. Δεν είναι ο σωστό τρόπο αυτό. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Το σημείωσαν ε, την, την ε, σοφή αυτή παρατήρηση του εισηγητή μα υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Ο εισηγητή μετά από όλε αυτέ τι διευκρινήσει συστήνει να υπερψηφίσουμε τη μεταφορά. Ποιοι είναι υπέρ, σα ευχαριστώ. Ποιοι είναι κατά, δύο. Σα ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν αποχέ. Εγκρίνεται. Je crois que nous avons épuisé les virements. Je crois que nous avons épuisé. Νομίζω πως εξαντλήσαμε την ημερήσια διάταξη τώρα. Επόμενη μας συνεδρίαση είναι στις 8 του μηνός. Στις 3. 3 ε, με 6.30. Και να σας ανακοινώσω από τώρα ότι η μεθεπόμενη δυστυχώς θα είναι πολύ καιρό μετά, μόνο στις 26 Ιανουαρίου. Προετοιμαστείτε ψυχολογικά. Αυτά, πέρα τη σα και καλή τύχη για την επιστροφή σας.